Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, επίσης, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για όλες τις ερωτήσεις σας και για την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή ιδεών που είχαμε σήμερα και σας διαβεβαιώ για ένα πράγμα. Αν τελικά με υποστηρίξετε και αν μου δείξετε εμπιστοσύνη, θα μετατρέψω τα λόγια μου σε δράση, σε πράξεις. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης προσπάθησα να σας δείξω ποια θα είναι αυτή η δράση που θα αναλάβω μαζί με εσά, με τα κράτη-μέλη και με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επενδύσει σε οικονομική ανάκαμψη και στην προώθηση της απασχόλησης. Θέλουμε να επιστρέψουν εκεί που θέλουν δουλειά σε θέσεις εργασίας, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να βελτιώσουμε την κινητικότητά τους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή κοινωνική προστασία και για τους εργαζόμενους ανθρώπους και τους μη εργαζομένους και θέλουμε να δεντικοποιήσουμε την μάχη κατά της ένδυας. Στόχος μας καλές και υγιείς συνθήκες εργασίας, θα καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ και άλλες καταχρήσεις και θα πολεμήσουμε για δίκαιες και ίσες δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η σαφής στόχη που έχουμε καθορίσει. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, θέλω να χρησιμοποιήσω πλήρως τα διαθέσιμα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσει μέχρι 300 δις ευρώ για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός μου αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού ευρωπαϊκού προπολογισμού Με αυτά τα χρήματα θα προσπαθήσω να πετύχω τους στόχους που ανέφερα, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να ενισχύσουμε την κοινωνική προστασία και να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Η εγγύηση για τους νέους θα είναι από τις βασικές μου προτεραιότητες και θέλω αυτό το μέσο να εφαρμοστεί πλήρως από όλα τα κράτη-μέλη χωρίς καθυστερήσεις. Στόχος μας προσμετρήσιμα αποτελέσματα διαρκείας. Η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική θα αποτελέσουν σαφέστερο, πιο ξεκάθαρο τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει. Θα κρυθούν βάσει των κοινωνικών του επιδόσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη φιλοδοξία να κινηθεί ενωμένη σαν ομάδα υπό την ηγεσία του Jean-Claude Juncker. Θα συνεργαστούμε και με το Κοινοβούλιο και βέβαια και με τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Κατανοούμε ότι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα και μπορούμε να πετύχουμε μόνο αν τα αντιμετωπίσουμε μαζί. Αν σε πέντε χρόνια μπορούμε να πούμε ότι σήμερα η Ευρώπη έχει περισσότερες απασχόλησεις, έχει λιγότερη φτώχεια, τότε θα ξέρουμε αγαπητοί συνάδελφοι και μόνο τότε θα γνωρίζουμε ότι πραγματικά κάναμε τη διαφορά για το λαό. Και όπως είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, για το λαό δημιουργούμε την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι για τους λαούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Once uh, Σας ευχαριστώ κυρία Τάισεν εκ νέου. Ευχαριστώ όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην υποβολή των ερωτήσεων. Η συνεδρίαση των συντονιστών θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών για να αξιολογήσουμε την ακρόαση από τις 1 μέχρι τις 2 στην ASP 5G2. Η συνεδρίαση των συντονιστών για την αξιολόγηση των ερωτήσεων και απαντήσεων 1 με 2 στην ASP 5G2. Σας ευχαριστώ όλους. Γεια σας.